Uh, Καλημέρα σας. Αρχίζουμε. Το πρώτο θέμα στη ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο στη Ρουμανία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου και το επόμενο θέμα αφορά τη Βουλγαρία στο ίδιο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου ο οποίος θεσπίστηκε μετά την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και λήψεις και δυναμίες στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και καταπολέμηση της διαφθοράς. Έκτοτε οι εκθέσεις αυτές προσπάθησαν να εστιάσουν στις προσπάθειες των αρχών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας με ειδικέ συστάσεις και έχουν καταγράψει και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η έκθεση του 2017 δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλέσαμε τον κύριο Williams από την ε, Γενική Γραμματεία ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, μας παρουσιάσει το θέμα αυτό και να γίνει συζήτηση με το μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Γουέλεμς Λύση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε και την Επιτροπή σας που δίνετε στην, την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας παρουσιάσουμε τις δύο εκθέσεις που εκρίναμε τον Ιανουάριο. Φέτος είναι κάπως διαφορετική η προσέγγιση των δύο εκθέσεων σε σχέση με το παρελθόν ε, κοιτάμε την πλήρη περίοδο που μεσολάβησε, τη δεκαετία από το 2007 μέχρι σήμερα και μας επιτρέπει αυτό να κάνουμε μια καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας και του μη αντιστρεπτού ε, των μεταρρυθμίσεων. Ε, έχουμε λοιπόν μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση φέτος και ελαφρώς διαφορετική δομή σε σχέση με το παρελθόν κοιτάξαμε την αρχική απόφαση για το μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου και τις ε, προσπάθειες που έχουν κάνει, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα. Είναι ενθαρρυντικά και παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή και η λειτουργία του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου. Κάναμε και πάρα πολύ συγκεκριμένε συστάσεις για το πώς θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Καμιά φορά στο παρελθόν Μαζί τους, να διευκρινίσουμε το πεδίο εφαρμογή και το τι θέλουμε να γίνει οι δύο χώρες. Οι εκθέσεις με τον τρόπο που έχουν πλέον διαρθρωθεί, σε αυτό αποσκοπούν ακριβώς να είναι πιο σαφείς οι συστάσεις, πιο πλήρεις, πιο οριστικές και τουλάχιστον όπως περιγράφεται στις εκθέσεις να μην ε, αντιστραφεί αυτή η πορεία η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Υπάρχουν κάποια ορόσημα για τη συγκριτική αξιολόγηση, κάποια benchmarks και ε, για το μέλλον κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και θα κλείσει αυτός ο μηχανισμός όταν θα έχει εκπληρώσει το σκοπό του και όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλες οι συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει να γίνει αυτό κατά τη διάρκεια της παρούσης θητής. Ωστόσο, για να ε, εξασφαλιστούν τα αποτελέσματα ε, και να είναι μόνιμα και βιώσιμα, χρειάζεται και συνεργασία και δέσμευση και προσήλωση στους στόχους αυτούς. Αναρωτήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν πραγματικά οι μηχανισμοί που επιτρέπουν ε, στα κράτη-μέλη να δείξουν ότι υπάρχει και η βούληση και η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη βιωσιμότητα. Και βεβαίω παρακολουθούμε και τι επιδόσεις και την απόδοση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίση να δράξει την ευκαιρία για να τονίσει και στις δύο εκθέσεις ότι δεν θεωρεί σκόπιμο να συνδέεται ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου με αποφάσει που λαμβάνονται σε άλλου τομεί. Ε, λοιπόν, αρχίζουμε από τη Βουλγαρία για να δούμε την έκθεση μία-μία. Πού μα οδήγησε η ανάλυση τη παρελθούση δεκαετία. Ε, Υπάρχουν διάφορες πτυχές ε, της ε, του δικαστικού συστήματος. Το πρώτο βήμα ήταν ένα σταθερό συνταγματικό πλαίσιο. Έγινε πρόοδος για το λοιπό νομικό πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το 2015 άρχισε η μεταρρυθμιστή δικαιοσύνης και παραμένει ένα βασικό στοιχείο με τις πρόσφατες ε, αλλαγές έχει δύο τμήματα το συνταγματικό δικαστήριο για να ασχολείται ε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς ε, είναι πιο διαφανής η λειτουργία και κάθε δικαστής έχει μία ψήφο για τις εκλογές. Και οι εκλογές του ε, θέρους θα είναι αποφασιστικές για να δούμε εάν εμπνέει το νέο σύστημα την εμπιστοσύνη τη κοινή γνώμη. Επίσης, οι δικαστές έχουν περισσότερο ε, λόγο και συμμετοχή στη διαχείριση των δικαστήριων. Και ο ποινικό κώδικα έχει αλλάξει και στη λειτουργία του και στη δομή του και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ε, η εισαγγελία και ε, διώκεται η διαφθορά. Το 2016 έγινε μια προσπάθεια που κατέληξε ε, σε μια ανεξάρτητη ε, ανάλυση και εκτίμηση ε, της βουλγαρικής εισαγγελία. Παραμένουν προβλήματα όμως και προκλήσεις στις ποινικέ διώξεις και στη δίωξη του σοβαρού εγκλήματος στην πάταξη τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αναγνωρίζει η έκθεση ότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές Στη Ρουμανία έρχομαι τώρα. Ενώ η Βουλγαρία έχει περίπου ευθυγραμμιστεί με τα άλλα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές αλλαγές υπάρχουν αδυναμίες, όπως είναι ε, στην ποινική δικαιοσύνη για παράδειγμα. Ε, άλλα προβλήματα και προκλήσεις που παραμένουν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες αμέσως μετά την ένταξη ε, των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια στρατηγική που ενέκρινε η Ρουμανία το 2015. Αυτή η στρατηγική είναι ακόμα στα σπάραγανα. Ε, και ο νόμος για την καταπολέμηση της διαφθοράς που κατατέθηκε η πρώτη φορά το 2015 δεν προχωράει ικανοποιητικά. Γιατί δεν υπάρχει και πολιτική συνένεση. Γιατί δεν τελεισιδικούν οι υποθέσεις στη Βουλγαρία κυρίως. Ε, Τη στρατηγική καταπολέμηση τη διαφθοράς το 2015 περιλαμβάνεται μια αποτελεσματική αρχή πάταξη της διαφθοράς, ε, όχι μόνο της υψηλής ε, διαφθορά, αλλά και τη χαμηλής καθημερινής σε τομεί υψηλού κινδύνου. Γενικώ, ε, πάντως για τη Βουλγαρία υπάρχει πρόοδο πλην όχι τόσο εντυπωσιακή όσο στην αρχή ή τόσο ταχεία και παραμένουν ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, οι συστάσεις μπορούν να επιτευχθούν στον χρονικό ορίζοντα που καλύπτεται την έκθεση. Τώρα έρχομαι στη Ρουμανία. Όλα αυτά ήταν για τη Βουλγαρία. κάναμε μια ανασκόπηση της δεκαετίας και διαπιστώσαμε σημαντική πρόοδο σε αρκετούς τομείς. Στη δικαιοσύνη υπήρχαν μεγάλες θεσμικές εξελίξεις. Αυξήθηκαν και οι πόροι στη δικαιοσύνη. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο καθιερώθηκε ως διαχειριστής του δικαστικού συστήματος και υπερασπιστής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα θέμα που έχει να κάνει με τη μη εκτέλεση των δικαστικών ε, αποφάσεων. Υπάρχουν ε, υπερβολικές επιθέσεις ε, και από τους πολιτικούς και από τα μέσα ενημέρωσης ε, εις βάρος δικαστών και Ε, Έχει γίνει προσπάθεια εξυγχρονισμού του αστικού και του ποινικού κώδικα για τη δίκαιη δίκη και για αποτελεσματικές διαδικασίες σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο. Είναι περιορισμένη λοιπόν ε, η έκταση για την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμών. Το νέο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που άρχισε να λειτουργεί φέτος θα έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ε, στην ε, στρατηγική των μεταρρυθμίσεων για την ακαιρεότητα. Υπάρχει ένας ε, εθνικός οργανισμός ακεραιότητας που έχει ε, προχωρήσει και έχει δώσει σημαντικά αποτελέσματα από το 2013 ακόμα και σε βέστους τομείς όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις ή εκλογές. Παραμένουν κάποια ερωτηματικά για το νομικό πλαίσιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά. Ακόμα δεν έχει ε, καθιερωθεί, δεν έχει θεσπιστεί ένα σαφές θεσμικό νομικό πλαίσιο που να εγγυάται τη βιωσιμότητα και την αηφορία. Επίσης υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την υλοποίηση ε, των ε, αποφάσεων του οργανισμού ε, αυτό, ακόμα και αν συνοδεύω από δικαστικές αποφάσεις. Ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου έχει διαπιστώσει μεγάλα προβλήματα διαφθορά, παρόλο που η χώρα έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Με το νέο οργανισμό που συστήθηκε και άρχισε να λειτουργεί, γίνει και άλλη πρόεδρος, παρόλα αυτά ε, δεν είναι σταθερό πάντα το νομικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο και αυτό το ε, σημειώνουμε στην έκθεση του Ιανουαρίου. Επίσης, οι ε, δικαστές ε, ε, υφίστανται μεγάλες επικρίσεις από το πολιτικό σύστημα και το μηντιακό σύστημα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ζητήματα άρσης ασυλίας ή άρνησης άρσης ασυλίας πολιτικών η δίωξη διαφθοράς υψηλού επίπεδου είναι προτεραιότητα πλέον ε, της εισαγγελίας στη Ρουμανία και η Εθνική Στρατηγική κατά της διαφθοράς παρέχει ένα σημαντικό θεσμικό πλαίσιο προς το σκοπό αυτό, ωστόσο χρειάζεται ακόμα να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια για την πρόληψη της διαφθοράς και με αποτρεπτικά μέτρα και στην δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει να κλείνουν τα παραθυράκια που ε, επιτρέπουν τη διαφθορά. Γενικώ ε, και συμπερασματικά. Οι δύο εκθέσεις ε, έχουν μια θετική αξιολόγηση για τις δύο χώρες και ε, εάν πληρωθούν όλες οι συστάσεις μπορεί τελικά και δικαιολογημένα να τερματιστεί ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου. Βεβαίως, εάν οι εξελίξεις ανατρέψουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αυτό αφορά κάποια βήματα που έκανε η Ρουμανία τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε τώρα οι κυβερνήσει των δύο κρατών μελών να επιτρέψουν την αγαστή συνεργασία όλων των θεσμών έτσι ώστε να ε, ε, εφαρμοστούν οι συστάσεις και να ολοκληρωθεί και να κλείσει ο μηχανισμός αυτός συνεργασίας και ελέγχου. Το πότε θα γίνει αυτό εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη όλων των ενεχομένων κυβέρνησης, δημόσιας διοίκησης, ε, άλλων φορέων, δικαστών κτλ. Ελπίζουμε αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα να παροτρύνει και να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις για να φτάσουμε σε αίσιο πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. The floor is now... Ευχαριστώ. Ο λόγος τους βουλευτές. Η κυρία Μακοβέη και Στέβενς Γραπίνη, Σόγκορ θέλουν τον λόγο. Ποιος άλλος θέλει τον λόγο. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ. So we start uh, in the order of the group and... Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε τις ομάδες, τις πολιτικές ομάδες με τη σειρά. Η κυρία Γκάμπριελ. Miss Gabriel, you have the floor. That's fine. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω βουλγαρικά. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του μηχανισμού. Δέκα χρόνια λοιπόν από την προσχώρηση των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και 10 χρόνια από την ε, καθιέρωση του μηχανισμού. Να πω λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμος για την δρομολόγηση των μεταρρυθμίσεων. Ο μηχανισμός βοήθησε την βουλιαρική κυβέρνηση στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη και στην μάχη κατά διαφθοράς. Να προσθέσω επίσης ότι προσφάτως πολλά ζητήματα προέκυψαν και ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, σαφή κριτήρια βάσει τα οποία κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι πρέπει να εγκατελευθεί ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός ε, είναι σημαντικός ως πλαίσιο, διότι θέτει προθεσμίες για την επίτευξη κάποιων στόχων αναφοράς. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Κομισιόν, διότι στην ε, πιο πρόσφατη έκθεση, την τελευταία έκθεση, ορίζονται και καταγράφονται τα βήματα τα οποία σημειώθηκαν, η πρόοδος που σημειώθηκε και μάλιστα για πρώτη φορά διατυπώνονται πολύ συγκεκριμένες συστάσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Στην περίπτωση που υλοποιηθούν αυτές οι προτάσει, συστάσει, Θα καταργηθεί ο μηχανισμός. Βλέπω για παράδειγμα συστάσεις όσον αφορά την διαφάνεια, την υποβολή τακτικών εκθέσεων κλπ. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Πώς θα γίνουν όλα αυτά εν τέλει. Θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία που ακολουθούσαμε ως σήμερα όσον αφορά το κράτος δικαίου για παράδειγμα κρίσιμο θέμα Εκεί είχαμε τακτικό διάλογο με την Κομισιόν. Τι ακριβώ θέλετε λοιπόν να αλλάξουμε. Και επειδή ανέφερα το κράτο δικαίου, να πω και πάλι ότι πέρσι τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόταση είναι έναν υποχρεωτικό ευρωπαϊκό μηχανισμό σχετικά με το κράτο δικαίου, που μάλιστα θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Ο μηχανισμός αυτός θα συμβάλλει στην συστηματική συγκριτική αξιολόγηση της πρόοδου όλων των χωρών και αποτελεί ένα ξεχωριστό μηχανισμό. Μήπω θέλω να πω ότι ο αντίστοιχο μηχανισμό που είναι ειδικό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πρέπει να εγκαταληφθεί. Για να δούμε πώ θα επιταχύνουμε λοιπόν την ε, πρόοδο και την υλοποίηση των συστάσεων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Κάποιοι από αυτούς δεν αφορούν τις δύο χώρες. Εννοώ ότι είναι θέματα στα οποία μπορούμε να κάνουμε πρόοδο όλοι μαζί. Κράτος δικαίου, διαφάνεια κλπ. Γι' αυτό ίσως και κάποιοι από τους μηχανισμούς που αφορούν συγκεκριμένα και μόνο κρατημέλη νομίζω πρέπει να αναθεωρηθούν. Διότι τα θέματα είναι κοινά. Χρειαζόμαστε κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό. Ας πούμε για την δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό εννοούσε νομίζω και ο κύριος Γιούνκερ όταν έλεγε για την ε, καταρρίξη αυτού του μηχανισμού εντός της παρούσας θητείας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Καπίνη. Ε, κυρία ευχαριστώ και εγώ θα μιλήσω ρουμανικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίαση. Εγώ θα αναφερθώ, όπως και συνάδελφος, ε, στα δύο κράτη. Μιλάμε για μία δεκαετή ανάλυση. Βλέπουμε την εξέλιξη στη Ρουμανία και χαίρομαι διότι έχουν καταγραφεί η πρόοδος και η πρόθεση πρόοδου. Όπως είπες και η συνάδελφος από το ΕΛΚ, μιλάμε για ένα μηχανισμό για δύο χώρες, ο οποίος είναι πλέον απαρχαιωμένος. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει ένας ε, εποπτικός μηχανισμός για τα 27 κράτη, γιατί η διαφθορά και η οικονομική πραγματικότητα είναι ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο και ίσως θα πρέπει να έχουμε μία χαρτογράφηση των 27 κρατών μελών. Θα ήθελα να πω Καταρχήν, ότι είπατε ότι το δικαστικό σύστημα ε, δεν είναι στο απειρόβλητο. Μπορείτε νομίζω να κρίνετε έναν εισαγγελέα, ένα δικαστή, όχι όμως το σύστημα στο σύνολό του. Το δικαστικό σύστημα λειτουργεί άψαχα, άψογα και αυτό το βλέπουμε γιατί υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός του δικαστικού από το 16 και μετά. Υπάρχουν ε, ορισμένα ολισθήματα τα οποία πρέπει να στυλιτευτούν, αλλά το σύστημα στο σύνολό του δεν είναι καθόλου κακό. Ποια είναι η προοπτική της ε, Επιτροπής, ποια είναι η οπτική γωνία μάλλον της Επιτροπής μετά από 10 χρόνια, τι προβλέπει. Δεν θα ήταν σκόπιμο να ε, προβάλετε μία μελέτη για ένα σύστημα ελέγχου για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ζήτησα να είναι υπόλογοι και οι δικαστές και οι δικαστικές αρχές στα 27 κράτη-μέλη με ένα νέο μηχανισμό και όχι αυτόν που είναι απαρχαιωμένος. Η κυρία Μακοβέ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απόφαση που έλαβε το Δεκέμβριο του 2016 να επιβάλλει μαζί με αυτές τις δύο χώρες από την 1η του 2017 να ε, εγκρίνουν ένα μηχανισμό ε, ελέγχου και επαλήθευσης και συνεργασίας, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Μιλάμε για το 15 και 16 και μιλώ για τη Ρουμανία, δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την καταπολέμηση της διαφθοράς σε αυτή τη διετία. Αν δούμε το, τους μηχανισμούς αυτούς συνεργασίας και ελέγχου τα τελευταία δέκα χρόνια βλέπουμε ότι όλοι συνεργάστηκαν. Έχουμε καταδικάσει και πολιτικούς από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, διάφορους μεγιστάνες, πολιτικούς, δικαστικούς. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό γιατί ο νόμος είναι ίσως για όλους και αυτό το είδαμε στην πράξη. Η Επιτροπή μίλησε για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Βλέπουμε όμως ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία και πολλές φορές καταδικάστηκαν πολιτικοί. Ε, εγώ έχω πει πολλές φορές σε σχέση με αυτό τον ελεγκτικό μηχανισμό ότι χωρίς αυτόν η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς δεν θα υπήρχε στη Ρουμανία. Ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου προβλέπει μεταξύ άλλων να συνεχίσει τη δραστηριότητα η δική μας αρχή δίωξης εγκλήματος και καταπολέμησης της διαφθοράς, η Δένεα και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ε, δραστηριοποίησης, δίωξης και πολιτικών προσώπων. Ο μηχανισμός ελέγχου και συνεργασίας θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι, μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι στόχοι. Και αυτό το συζητήσαμε και με άλλους συναδέλφους, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό ελέγχου και συνεργασίας σε επίπεδο όλων των κρατών μελών. Να προβλέπεται ένας τέτοιος ε, μηχανισμός ε, λογοδοσίας. Όσο περισσότεροι μηχανισμοί υπάρχουν, τόσο περισσότερη πίεση υπάρχει κατά των πολιτικών έτσι ώστε να διώξουν το έγκλημα και τη διαφθορά γιατί ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλές ε, καταχρήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, καταδικάστηκαν πολιτικοί από την ανεξάρτητη δικαστική αρχή στη Ρουμανία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις δημόσιες προμήθειες, γιατί και εκεί υπάρχει διαφθορά. Για τη Ρουμανία θα πρέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα και σε εσωτερικό επίπεδο, δηλαδή θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, θα μεταρρυθμίσουμε το δικαιοδοτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να έχουμε μία εύρωστη δημοκρατία. η διαφθόρα δεν επιτρέπει να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός και εμπιστοσύνη στον κρατικό μηχανισμό. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πιστεύω ότι όσο περισσότεροι μηχανισμοί υπάρχουν τόσο το καλύτερο γιατί έτσι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση κατά των πολιτικών που δεν είναι συνεργάσιμοι. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Χουισμένοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Επιτροπή μας εδώ συζητούμε μία από τις πολλές επιτροπές για τον Μηχανισμό Συνεργασίας και Ελέγχου για την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Τι αλλάζει όμως σήμερα. Η αναχείρας έκθεση προβαίνει σε διαπιστώσεις και δείχνει τον δρόμο προς τα εμπρός. Πολλές φορές συζητήσαμε στην Επιτροπή μας εδώ κάποιες ε, δυσαρμονίες, ε, ασυνέπειες των εκθέσεων κλπ. Όμως, η έκθεση λέει σήμερα ότι ακολουθώντας τις συστάσεις, οι χώρες, οι δύο χώρες μπορούν να πετύχουν τους στόχους αναφοράς, ακολουθώντας τις συστάσεις. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το κράτος δικαίου. Η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα και δεν νομίζω ότι αυτές οι στάσεις μπορούν να ή πρέπει να εφαρμόζονται εκεί και ω έτυχεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σημειώνει ότι οι δύο χώρες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ικανοποιούν όσον αφορά την δικαιοσύνη και όμως παρόλα αυτά ο μηχανισμός εργασία και ελέγχου συνεχίζει να ισχύει για τις δύο αυτές χώρε και μόνο, όχι όμως για τι άλλε χώρε μέλη. Το βρίσκω αυτό κατά και η βάρο των δύο χωρών μας στο πλαίσιο του Σέγγεν. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των συμπερασμάτων του μηχανισμού ε, με άλλες πολιτικές, μεταξύ άλλων και το Σέγγεν. Η έκθεση, δυστυχώς, χρησιμοποιείται για να κρατούνται αυτές οι δύο χώρες εκτός Σέγγεν, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλα κριτήρια. Ελπίζω λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα αντικατασταθεί από ένα κοινό μηχανισμό που θα ισχύει για όλες τις χώρες και όχι μόνο για τις δύο συγκεκριμένε. χάρη στον οποίο να γίνουν και αλλαγέ με τρόπο διαρκή και βιώσιμο. Αυτό το τονίζω. Ο μηχανισμός πρέπει να αφορά όλα τα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Ο Thank e Με την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ρουμανία έχει κάνει μεγάλες προόδους στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και ελπίζω αυτό να μην σταματήσει στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, 10 χρόνια μετά την ένταξή της, είναι τελευταία ουραγός η ε, Ρουμανία ε, στις επιδόσεις ε, της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί σημαντικές ανησυχίες για τις δικονομικές εγγυήσεις, για τα στάδια της δικαιοσύνης και παραβιάσεις στοιχειωδών κανόνων του κράτους δικαίου. ο ε, ε, ε, οργανισμός DNA του 2015 έχει ερευνήσει ένα σχολείο που ιδρύθηκε από την Καθολική Εκκλησία και που φοιτούν 400 παιδιά. αυτά είναι ανεφροηγουμένα που συμβαίνουν στη Ρωμανία, προς τις διώξεις και το δικαστικό σύστημα. Ε, μπορεί να έχουν γίνει πρόοδοι, αλλά παραμένουν ακόμα ε, μεγάλα προβλήματα και δεν τα έχει αντιμετωπίσει ακόμα ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου. Οι εθνικές μειονότητες ε, το έχουν ξαναζήσει αυτό. Μόλις χαλαρώσει η πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η, πρόεδρος, πρόοδος που έχει επιτευχθεί μπορεί να καταστραφεί. Δεν εφαρμόζεται ε, στην πράξη νομοθεσία ακόμα ε, παρεμποδίζονται ορισμένοι να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα καθώς επίσης και οι περιουσίες που επιστράφησαν μετά την αλλαγή του καθεστώτος ε, κατάσχονται ξανά από το κράτος. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για λήξη του μηχανισμού αυτού. Αντί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεσή τους. Ε, κοιτάξτε, θα πρέπει να θυμηθούμε την κατάσταση ε, που επικρατούσε όταν εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σε αντίθεση με κάποια άλλα νέα κράτη-μέλη, στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία βρήκαμε την εξής κατάσταση. Και οι δύο ήταν συγκρίσιμες με άλλες φτωχές χώρες, αλλά και στις δύο χώρες είδαμε ψηλά επίπεδα διαφθορά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, που δυστυχώς αυτό ήταν η κανονικότητα, η καθημερινότητα στη χώρα αυτή και στις δύο χώρες για πάρα πολλά χρόνια. Η προθυμία λοιπόν να αλλάξει αυτό εκδηλώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δύο αυτές χώρες, εξού και ο μηχανισμός. Και Χαίρομαι που μετά από δέκα χρόνια που μια γενική θεώρηση στην ιστορία δεν είναι μεγάλη περίοδος, έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφύγουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει ε, επιτευχθεί πρόοδο στη δικαιοσύνη και στην ε, επιβολή του νόμου. Ε, ε, πρόοδος μεν πλην αργή. Αυτό παρατηρείται όμως και σε άλλα κράτη-μέλη και διαφθορά και ε, ε, ζητήματα που ε, έχουν να κάνουν με τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα, εκεί η πρόοδος είναι αργή. Δεν είναι μόνο η Βουλγαρία και η Ρουμανία, έχει αλλάξει κατάσταση και σε άλλα κράτη-μέλη και με αργούς ρυθμούς και θα ήθελα να ακούσω και άλλους συναδέλφους που επανειλημμένα κατηγορούν τη Ρουμανία θα πρέπει κατά τον ίδιο τρόπο ας πούμε, να αναφερθούμε δυστυχώ και στην Ουγγαρία, όπου και διαφθορά υπάρχει και ε, κακοδιαχείριση ε, του δημοσίου χρήματος, έχουμε εκθέσει τη Όλαφ και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε αυτό για πολιτικά παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλες χώρες λοιπόν με φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και σε λεγόμενες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό Χαίρομαι ε, που έχουμε αυτό το μηχανισμό, χαίρομαι που έχει επιτευχθεί η μεγάλη πρόοδος και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και τις δύο χώρες, και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Εγώ δεν βλέπω προθυμία, ούτε μειωμένη διάθεση. Βεβαίως χρειάζεται υποστήριξη. Δυστυχώς αυτό που χρειάζεται και συμφωνώ με κάποιους συναδέλφους είναι να έχουμε αντίστοιχους μηχανισμούς ε, και ε, πίεση σε σχέση με τις εξελίξεις σε κάποιες άλλες χώρες και δεν θα πρέπει να εθελοτυφλούμε απέναντι σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, the next is... Επόμενη η κυρία Χέλγα Στέβενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκθέσεις για το μηχανισμό ελέγχου και συνεργασίας. Η Ρουμανία σημείωσε σημαντική πρόοδο και πρέπει να συνεχίσει στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Για να συνεχίσει ο αγώνας να είναι ποιοτικός, ο μηχανισμός ε, και ο οργανισμός κατά της ε, διαφθοράς και οι άλλοι φορείς πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, να μην αλλάξει η διαδικασία ορισμού εισαγγελέων και άλλων υπευθύνων. Η υπηρεσία, η DNA και οι εισαγγελείς πρέπει να διορίζονται με βάση τον υφιστάμενο μηχανισμό ο οποίος έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του. Δεν χρειάζονται λοιπόν αλλαγές εκεί, ούτε στο νομικό πλαίσιο της ε, Εθνικής Διεύθυνσης κατά της διαφθοράς στη Ρουμανία, ο αγώνα κατά τη διαφθορά, έχει σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν ε, βλέπω γιατί λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού που αποδίδει τόσο καλά. Να σταματήσουμε ίσα ίσα να περιορίζουμε τις αρμοδιότητε αυτού του οργανισμού. Ίσα ίσα πρέπει να ενισχύσουμε τον, την ε, DNA και του εγγελείς που μάχονται κατά τη διαφθορά. Ο μηχανισμό εργασία και ελέγχου και η Κομισιόν πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ε, Ρουμανία στον αγώνα κατά τη διαφθορά. Δεν είναι δυνατόν να μεταχειριζόμεθα την Ρουμανία σαν δε, ε, χώρα δεύτερη κατηγορία. Και το ίδιο ισχύει για του πολιτικού τη. Άλλωστε, γι' αυτό η Ρουμανία είναι στην Ευρώπη και η Ευρώπη συμπεριλαμβάνει τη Ρουμανία. Υπενθυμίζω ότι το κράτος δικαίου αποτελεί μία από τι θεμελιώδει αρχέ λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφθορά σκοτώνει, η διαφθορά έχει θύματα σε όλα τα επίπεδα, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, στους δημόσιους θεσμούς και στα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Ράντεν. Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την έκθεση. Εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία θα έλεγα ότι πριν από 10 χρόνια προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τότε έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και στον αγώνα κατά της διαφθοράς, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στην έκθεση του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου. Οι εκθέσεις όμως δεν οφείλονται στον μηχανισμό, αλλά στην βούληση του βουλγαρικού λαού για δικαιοσύνη και για λιγότερη διαφθορά. Στη Βουλγαρία προσπάθησαν και τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία να γίνουν πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά στον αγώνα κατά της διαφθορά Αυτό περιμένει και ο βουλγαρικός λαός. Τα συμπέρασματα στην έκθεση δεν διατυπώνονται με τρόπο συστηματικό. Υπάρχουν ασυνέπειες, ε, ούτε βεβαίω ε, αποτελούν Ευαγγέλιο. Από τους πέντε που συνέταξαν την έκθεση, δύο μόνο είναι πλήρους απασχόληση στον τομέα και πολύ λίγοι έχουν πείρα με θέματα δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να παρακολουθήσουν τι μεταρρυθμίσει στη δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, οι μεταρρυθμίσει στη δικαιοσύνη συνεχίζονται. Συνεχίζονται επειδή το θέλουμε, όχι επειδή μα το πάνε αλλά διότι, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο προσμένει η κοινωνία των πολιτών στη Βουλγαρία. Είναι κάτι το οποίο ζητάει η χώρα μα, ο βουλγαρικό λαό. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε βεβαίω με την προσχώρηση των δύο χωρών. Σήμερα όμω αυτό ο μηχανισμό δεν είναι πλέον αποτελεσματικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι αποτελεί και διάκριση βάρο των δύο χωρών, διότι ισχύει και λειτουργεί μόνο για τις δύο συγκεκριμένε χώρες. Τη στιγμή μάλιστα που ξέρουμε ότι η διαφθορά υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ, ο μηχανισμός αυτός γίνεται αντικείμενο κατάχρηση για πολιτικού σκοπού. και εν τέλει απαγορεύει την συμμετοχή των δύο χωρών στο Σέγγεν. Παρά το ότι δεν αποτελεί επίσημη απέτηση για συμμετοχή στο Σέγγεν. Οι επενδύσει λοιπόν όσον αφορά τη δημοκρατία πρέπει να σταθμίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία μάλιστα θα ισχύουν με τον ίδιο ακριβώ τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Εν κατακλείδη θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν πόσο κοστίζει πραγματικά να εκπονηθεί μια τέτοια έκθεση από τον μηχανισμό. Πόσο κοστίζει για τον, ευρωπαϊκό, για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Διότι όλα αυτά ανατίθενται σε εξωτερικού συνεργάτε, εμπειρογνώμονε κλπ. Πόσα πληρώνουμε τόσα χρόνια. Το θέμα είναι να έχουμε λοιπόν έναν πανευρωπαϊκό μηχανισμό για όλες τις χώρες και όχι μόνο για τις δύο. Επόμενο ομιλητή και τελευταίος ομιλητή στον κατάλογο μου είναι ο κ. Παύλ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω την πρόοδο στην οποία αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το μηχανισμό ελέγχου και συνεργασίας στη Ρουμανία τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει. Πρόκειται για έναν μηχανισμό ο οποίος ισχύει για μόνο αυτά τα δύο κράτη, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο ο κύριος Τίμερμανς, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μαζί με τον Πρωθυπουργό Γκριντεάνου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Τούτορ Τόντερ, μίλησε για πολύ θετικά βήματα στη Ρουμανία, η οποία ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη. Σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκαν. Μπορέσαμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αρθεί αυτός ο μηχανισμός άμεσα. Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση και από, το, από τη Ρουμανική Βουλή σχετικά με αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε ποια μέτρα θα ληφθούν έτσι ώστε να ε, αρθεί αυτός ο μηχανισμός, όταν πληρούνται βέβαια οι όροι. Αυτό αφορά και την ε, πρόσβαση, προσχώρηση στο χώρο Σέγγεν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο μηχανισμός, όπως και ο μηχανισμός του χώρου Σέγγεν, και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη στο δικαστικό τομέα στη Ρουμανία Πιστεύω ότι το κράτος δικαίου σημαίνει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να τηρηθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις χώρες και στη Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Um, Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάρκο το λόγο σύντομα, όμως ε, γιατί θα πρέπει να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Επειδή έγινε αυτή η διασύνδεση μεταξύ μηχανισμού και Σέγγεν, δεν το έκανα εγώ, αλλά το έκαναν οι συνάδελφοι, συνάδελφοι από άλλα ε, πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα οι σοσιαλιστές, θα ήθελα να πω τα εξής. Η Ολλανδία ήταν από τις χώρες ε, που είπε ότι θα ήθελε να προσχωρήσει η Ρουμανία στο χώρο Σέγγεν μετά από δύο εκθέσεις. Η πρώτη είχε συνταχθεί. Όμως η έκθεση που συντάχθηκε το 2012 έδειξε ότι δύο πολιτικά κόμματα ε, έχουν παραβιάσει το νόμο. Θυμόσαστε ακριβώς τι είχε γίνει τότε, το 2012, και δυστυχώς δεν ίσχυσε το κράτος, δεν υπήρχε κράτος δικαίου. Και γι' αυτό δεν μπήκαμε στο χώρο Χέγγεν. Δηλαδή το ΠΣΔ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και άλλα ήταν εκείνα που παραβίασαν το κράτος δικαίου. Okay. Um, yes. We Καλώς. Ας μην ξανανοίξουμε τώρα τη συζήτηση να την επεκτείνουμε σε άλλα θέματα, να περιοριστούμε στι εκθέσει για το μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου. Όλε οι πολιτικέ ομάδε έκαναν και σχόλια και ερωτήσει και γι' αυτό θα παρακαλούσα τώρα τον κύριο Σλέιζ, ε, τη Γενική Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα απαντήσει και να σχολιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και πάλι. Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω καλύπτοντας όλα τα θέματα που γραμμίζω πρώτα απ' όλα και θέλω να πω ότι αυτό με τη σημερινή σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι ακόμα σαφέστερο ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο κράτος δικαίου. Είναι θέμα το οποίο μας είναι ιδιαίτερος προσφυλές και όλοι οι ο κ έχει συμμετάσχει το περασμένο φθινόπωρο σε αυτήν την συζήτηση. Το ζητούμενο είναι ένας οριζόντιος ε, μηχανισμός για όλα τα κρατημέλη. Είναι θέμα, επαναλαμβάνω, το οποίο η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βλέπει ως θέμα το οποίο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύνολο της. πρέπει να καθιερώσουμε μηχανισμούς προς αυτήν την κατεύθυνση για το κράτος δικαίου δηλαδή ανεξαρτήτως των ε, εκκρεμών ζητημάτων επί των οποίων δεν έχει ακόμη καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι το θέμα του κράτους δικαίου είναι θέμα ιδιαίτερως προσφυλές ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το βλέπουμε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και για συγκεκριμένε περιπτώσεις και θέματα βάσει του πλαισίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το οποίο έχει διαμορφωθεί και στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχουμε μια ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσουμε τη δικαιοσύνη μας. Έτσι ώστε οι υποθέσεις που προκύπτουν να μπορούν να πάνε εν ανάγκη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωματών του Ανθρώπου. Ο μηχανισμός λοιπόν συνεργασίας και ελέγχου ας θυμόμαστε ότι προέκυψε λόγω συγκεκριμένων καταστάσεων αυτή τη στιγμή είναι υπό αναθεώρηση ως τμήμα ενός πλήθους άλλων ε, μηχανισμών με διαφορετικούς σκοπούς και όντως βεβαίω εστιάζεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Είναι όμως παράλληλα ένας μηχανισμός ο οποίος ε, δεν αποσκοπεί στην <laughs> τελειότητα αλλά σε ένα εύλογο επίπεδο επιδόσεων. Θα θυμάστε ότι για την Ρουμανία και τη Βουλγαρία τέθηκαν στόχοι θεωρήθηκε ότι η επιτεύξη του 70% ήδη θεωρήθηκε εύλογη και από τις δύο χώρες. Αυτό είναι λίγο πολύ και το επίπεδο το οποίο θέλει να πετύχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τον μηχανισμό πολύ σοβαρά Κάποιοι θεωρούν ότι δίνουμε υπερβολικά πολύ σημασία, αλλά το αντίθετο, το ίδιο και με τη συζήτηση περί των διερθεμένων πόρων. Εμεί πιστεύουμε ότι αφιερώνουμε στον μηχανισμό όσου πόρου απλώ απαιτούνται για να μπορέσει ο μηχανισμό να διεκπαιρεώσει τον ρόλο του με τρόπο εύλογο και αποτελεσματικό. Ακούμε φυσικά και τους άλλους δείτε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου από έτος σε έτος. Βλέπετε ότι η προσέγγιση μας, η μεθοδός μας αναπροσαρμόζεται, ενημερώνεται και γι' αυτό και δεχόμεθα και εύσημα κάθε χρόνο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο μηχανισμός προσφέρει υπηρεσία στα κράτη-μέλη με τρόπο που νομιμοποιεί θα έλεγα την ευρωπαϊκή διάσταση του πράγματος. Έχω συνεπώς την πεποίθηση ότι φέρνουμε σε πέρας τον ρόλο μας με τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο. Χάρηκα που άκουσα, πρέπει να πω, ότι υπέπεσε στην προσοχή των βουλευτών ότι διατυπώθηκαν και συγκεκριμένες συστάσεις. Μάλιστα τέθηκε το ερώτημα με ποιο τρόπο υλοποιούνται οι συστάσεις. Είναι μετά και το θέμα της υποβολής των εκθέσεων ε, και το θέμα δεν είναι μόνο τι στέλνεται στην Κομισιόν, το θέμα είναι τι ανακοινώνεται και προς τα έξω. Γιατί αυτό είναι, θα έλεγα, θεμέλιο για την βιωσιμότητα του συστήματος, για την η υπευθυνότητα όλων, τη λογοδοσία, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η σχετική πρόοδο σημαίνει με τρόπο, όπως είπα, βιώσιμο και διαρκή στις δύο συγκεκριμένε χώρες, ανεξάρτητα των όσων συμβαίνουν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για όλες τις εξηγήσεις που δώσατε και τις απαντήσεις. Ολοκληρώνονται τα δύο αυτά θέματα εδώ. Ευχαριστούμε και τους ομιλητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, το επόμενο σημείο στη διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντική πρόταση στην τρέχουσα μεταρρύθμιση του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Είναι η πρόταση, η οδηγία για τις απαιτήσει να γίνει κανονισμός. Η οδηγία αυτή είναι το εργαλείο με το οποίο συνδέεται και ενσωματώνει τη Σύμβαση Γενέβης για το καθεστώς του πρόσφυγα το 1951 στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Σημαντικός πυλώνας του συστήματος, η οδηγία ήδη αναθεωρήθηκε το 2011 και τώρα αλλάζει ε, το κείμενο, το νομοθέτημα και από οδηγία γίνεται κανονισμός, άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εναρμονίσει έτσι περαιτέρω τους κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την αναγνώριση των υπηκών τρίτων χωρών και των απατρίδων ως δικαιούχων δικαιού διεθνούς προστασίας. Επίσης, ορίζονται πρότυπα για τα δικαιώματα που ε, συνδέονται με το καθεστώς αυτό. Η κυρία Φαγιόν είναι η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Κατέθεσε την πρότασή της στις 9 Μαρτίου 2017 το σχέδιο έκθεσης και σήμερα θα συζητήσουμε τις 703 τροπολογίες που κατατέθηκαν εκτός των 95 της εισηγήτριας για τη διαδικασία αναδιατύπωσης. Θα δώσω πρώτο το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στους σκιώδεις. Καθίστε παρακαλώ. The Για να δώσουμε τη δέωσα προσοχή στην εισηγήτρια. Could you please sit down or take the talks outside of the room? Παρακαλώ καθίστε ή αποχωρήστε. Η κυρία Φαγιάννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω εδώ παρόντες όλους τους σκιώδεις ηγητές. Μάλλον συζήτηση με σκιώδης θα γίνει, αλλά την με αυτή τη συζήτηση, συνεδρίαση με τους σκιώδης ηγητές. Όπως είπατε κι εσείς, η έκθεση αυτή θέτει τα κριτήρια για τη διεθνή προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι αρκετά σημαντική. Όπως είπατε και εσείς, μαζί με τις δικές μου τροπολογίες, ε, οι υπόλοιπες τροπολογίες υπερβαίνουν τις 800 επί της προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον κανονισμό αυτό. Τέσσερις συνεδριάσεις κάναμε τους και οδησηγητές και ανταλλάξαμε ε, απόψεις, όπως και προηγουμένως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες και την κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους και και προσβλέπω και τη μελλοντική συνεργασία μας με όλους τους συναδέλφους. Ήδη έχουμε ε, αρχίσει να ε, συζητούμε για τις συμβαστικές τροπολογίες και χαίρομαι που στις τροπολογίες ε, αντικατοπτρίζονται πολλά από τα θετικά που ανέφερα και εγώ στο σχέδιο έκθεσης. Σε αυτό το πνεύμα θα συνεχίσω για τις συμβαστικές τροπολογίες. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, που προτείνει να βελτιωθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το κείμενο για τη διεθνή προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η κεντρική ιδέα για μένα. Να έχουμε μια πάρα πολύ ευρεία πλειοψηφία όσο γίνεται μεγαλύτερη για τις συμβαστικές τροπολογίες παρά το γεγονός ότι Υπάρχουν και κάποιες πάρα πολύ ακραίες θέσεις που εκφράζονται στις τροπολογίες από διάφορους συναδέλφους. Φαντάζομαι όμως θα βρούμε μια χρυσή τομή. Με χαράξα τους συναδέλφους και ό,τι σε προηγούμενες συνεδριάσεις να έχουν μια θετική ε, αντιμετώπιση για κάποια πάρα πολύ κρίσιμα για μένα και σημαντικά σημεία της έκθεσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός είναι από ε, τις πιο σημαντικές προτάσεις για το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και θα αντιμετωπίσει τα βασικότερα ε, θέματα που αναφέρω και εγώ στην έκθεσή μου. Ποια είναι αυτά θα πρέπει να δίνεται προστασία σε εκείνους που πραγματικά τη χρειάζονται για να έχουν την ευκαιρία να ξαναρχίσουν μια νέα ζωή με ε, αξιοπρέπεια, με ευημερία και με ασφάλεια κυρίως για ένταξη, ενσωμάτωση στη χώρα, ασφάλεια εργασιακή και ε, βεβαίως ε, και με τη δυνατότητα μετακινήσεων. προσπάθησα να πλησιάσω το καθεστώς του πρόσφυγα και εκείνου που έχουν δευτερογενή ε, προστασία ε, και να μειωθεί και ε, το διοικητικό και γραφειοκρατικό άκθος για τα κράτη-μέλη. αν δεν καταφέρουμε να εναρμονίσουμε το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάσουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα είναι κρίμα. Και είδαμε ε, τι έγινε με τις τελευταίες μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη. Μια από τις μεγάλες αλλαγές που προτείνεται στο σχέδιο έκθεσης είναι η διάρκεια των αδειών παραμονής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώ επέλεξε την εύκολη λύση και θέλησε να μην προτείνει βελτιώσεις. Εγώ διαφωνώ ε, Ξέρω ότι διαφέρουν οι πρακτικέ στα διάφορα κράτη-μέλη και επίση καταλαβαίνω τη θέση ορισμένων συναδέλφων, αλλά είμαι πεπισμένη ότι εμεί θα πρέπει να στοχεύουμε στο καλύτερο. Δηλαδή, μια πενταετία για την πρώτη παραμονή και μετά από την πρώτη πενταετία οι άνθρωποι που προστατεύονται από τη διεθνή προστασία ε, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και και να ε, έχουν παρατεταμένη ε, παραμονή ακόμα και ηθαγένεια. θα πρέπει για όλους αυτούς τους λόγους να ε, είναι κανονισμό στο κείμενο και όχι να επιστρέψουμε στην οδηγία γιατί η οδηγία παρέχει μια ευελιξία η οποία τελικά θα είναι εις βάρος του στόχου ε, της ε, πρότασης. Εμείς θα πρέπει να ε, έχουμε φιλόδοξους στόχους και να ζητούμε περισσότερο, όχι λιγότερο. Τώρα θέλω να ακούσω τους συναδέλφους. Ε, ολοκληρώνουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία και διαφορετικές απόψεις με στόχο να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας η έκθεση αυτή μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαγιόν. Ας ακούσουμε τους σκιώδεις τώρα. Για το ΕΛΚ. και η κυρία Μουσολίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα απαντήσω άμεσα στο θέμα αυτό, γιατί εμείς είχαμε πολλές επαφές και πολλά κοινά σημεία σε σχέση με την διατύπωση. Ε, για να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία καταρχήν και φυσικά να υπάρχουν μεγαλύτερη έλεγχη και ασφάλεια. Όπως ως προς το πρώτο σημείο της εισηγήτριας, θεωρούμε και εμείς ότι θα πρέπει να αρθούν όλα τα γραφειοκρατικά προσκόμματα χωρίς να υπάρχει παρανομία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, νομιμοποίηση και επικουρική προστασία για πέντε χρόνια. Συμφωνούμε δηλαδή με την πενταετία και επίσης ότι δεν θα πρέπει να επαναξε... επανεξεταστεί το καθεστώς τους ε, τη στιγμή που ζητάνε ε, ανανέωση άδειας ε, παραμονής. Δεν θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος πάλι από την αρχή, γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια για τους ανθρώπους αυτούς ιδιαίτερα αν πρόκειται για πάτριδες. Και ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου αλλάζει τις προδιαγραφές σε σχέση με τη χώρα προέλευσης. Όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να υπάρχει επικουρική προστασία, αλλά είμαστε υπέρ της αναλογικότητας, δηλαδή να δούμε αναπερίπτωση το ζήτημα σε σχέση με τη διεθνή προστασία και να μην επιβάλλουμε μια κύρωση που μηδενίζει το μετρητή σε σχέση με την πενταετία. Σε σχέση με την εσωτερική προστασία, θα πρέπει να είναι ε, όχι δεσμευτική, δηλαδή να ισχύει σε θελούσια βάση. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το κατά πόσο ετών ζητά διεθνή προστασία. Διαφορετικά τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες, δηλαδή μιλάμε για εσωτερική προστασία αλλά εάν δεν υπάρχει διμερή συμφωνία με τον λόγο κράτος μέλος, τότε υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία. Ως προς τους ανηλίκους, πάλι σε αυτό το θέμα, αυτό που έχει σημασία είναι οι πέντε ημέρες μη εργάσιμες, μη εργάσιμες, το τονίζω αυτό, και φυσικά να υπάρχει έλεγχος και να μην περνάει από ε, ίδρυμα σε ίδρυμα γιατί αυτό είναι πολύ αρνητικό για την ευάλωτη αυτή κατηγορία των ανηλίκων. Ευχαριστώ. Ε, η Ιούσι Χάλα από, τους, από το ECR. θεωρούμε ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε περαιτέρω τη διαδικασία χορήγησης ασύλου από πλευράς ECR, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για διεθνή προστασία σε πολίτες από τρίτες χώρες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός. Θα ήταν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ώστε η έκβαση της ε, διαδικασίας χορήγησης ασύλου να ε, μη σχετίζεται με το κράτος μέλος το οποίο ισχύει αυτή η προστασία. Θα πρέπει όμως το σύστημα χορήγησης ασύλου να μην ε, επιδοτεί την, τους οικονομικούς μετανάστες. Θα πρέπει βεβαίως να δίνονται ευκαιρίες και να μην υπάρχει διαδικασία δίωξης. Τα συστήματα ασύλου έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους που υφίστανται δίωξη, όχι όμως ε, να οθεί και να επικροτεί την ελεύθερη ροή μεταναστών από άλλες χώρες όπως ορίζουν και λένε οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές και αριστεροί. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε περισσότερη μετανάστευση στην οποία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά και κοινωνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής προστασία έχει πάντα προσωρινό χαρακτήρα. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν όταν δεν υπάρχει πια ανάγκη προστασίας. Φυσικά αυτός που ήρθε ως πρόσφυγας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ε, για χορήγηση διαμονής, εάν αυτός ή εκείνοι έχουν μπορέσει να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη μόνιμη διαμονή και στη χορήγηση υπηκότητας, ιδιαίτερα εάν οι, τα φυσικά αυτά πρόσωπα, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην τοπική κοινωνία. Έχουμε υποβάλει ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών που αντικατοπτρίζει αυτή τη, αντικατοπτρίζουν αυτή την πολιτική θέση. Ελπίζω να τις υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Για παράδειγμα, η διεθνής προστασία θα πρέπει να χορηγείται για ένα χρόνο κάθε φορά. Η ανάγκη προστασίας θα πρέπει να αποτιμάται κάθε φορά που ανανεώνεται η άδεια παραμονής. Γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει διοικητικό φόρτο, αλλά αυτό ε, σχετίζεται και με την παρουσία των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί και δεν μπορούν να παραμείνουν στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των μεταναστών και πιστεύω ότι ένας δικαιούχος χορήγησης προστασίας έχει και δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Δηλαδή η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση θα πρέπει να είναι πρόκριμα για να μπορέσει να ενσωματωθεί ο μετανάστης στη χώρα. Αυτό αφορά και την εκμάθηση της γλώσσας. Και θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος χωρίς άδεια όσοι προέρχονται από τρίτες χώρες δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες εάν έχουν ε, προβεί σε βίες πράξεις ή εάν έχουν παραπλανήσει και βιαιοπραγήσει κατά ανηλίκων ή εάν είναι ύποπτοι για τρομοκρατικές πράξεις. Θεωρώ ότι Μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες όταν μιλάμε για προστασία και ιδιαίτερα για διεθνή προστασία, αλλά δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, γιατί θεωρώ ότι να δεχόμαστε ακατάπαυστα ε, μετανάστες δεν δείχνει αξία, πραγματικές αξίες, αλλά ανευθυνότητα. Ευχαριστώ. Αγγελικά, από τους ελεύθερους ισχυώδες δεν είναι εδώ από ό,τι φαίνεται, οπότε συνεχίζουμε με αγκούα. Κύριε Βερζιά. Πρόεδρε, αντικαθιστώ την Μπάρμπαρα Σπινέλη, τη συναδελφό μου, η οποία ζητά την κατανόησή σα ε, για την απουσία της. Μου έστειλε όμως τα σχόλιά της, τα οποία θα προσπαθήσω να σας ε, καταθέσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν Σκιώδης για το εξαιρετικό έργο καταρχάς για την ε, λεπτομερέστατη ανάλυση είναι κατά τη, του επανακαθορισμού ή της τροποποίησης της αρχής της μη επαναπρόθεσης Διαφωνεί λοιπόν με τις προτάσεις του κανονισμού. Ήδη κατέθεσε αριθμό τροπολογιών που συνάδουν και υποστηρίζουν την αρχή της μη επαναπρόθεσης για να αποφύγουμε κάποιες παγίδες που ελοχεύουν στον κανονισμό έτσι όπως έχει δημορφωθεί από την Κομισιόν. Αυτά έχουν ως εξή. Καταρχήν, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο ορισμό, καλύτερη αναγνώριση αν θέλετε, ε, των περιβαλλοντικών προκλήσεων των μεταναστών. Έχουμε τους περιβαλλοντικούς πρόσφυγες και να προσθέσω προσωπικά ότι υπάρχουν τριπλάσια ιστορικώς εκτοπισμένοι στο ιστορικό δηλαδή χωρών σε σχέση με τους πρόσφυγες που μεταβαίνουν σε άλλη χώρα. Θέλω να πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ανθρωπογενή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις της, την ε, εκμετάλλευση, που προέρχεται από την ε, γεωργία και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητε, Μεταξύ άλλων και την ε, μαζική αρπαγή γεών. Για την επικορική λοιπόν τώρα προστασία και την αναγνώριση αυτών των ε, προσφύγων πρέπει να βασιστούμε στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάποια κρατημέλη. Η σκιώδης ισηγητρία επιθυμεί να οριστούν τα μέλη της οικογένειας ώστε να διευρυνθεί ο ορισμός της επανένωσης των οικογενειών για να ληφθούν υπόψη και οι οικογένειες έτσι όπως διαμορφώνονται μετά από την αύξηση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επίσης να καταργηθεί η υποχρέωση των κρατών μελών να παρακαθορίζουν μόνο τους το καθεστώς διεθνούς προστασίας οι έξι μήνες να γίνουν εννέα για να μπορούν να ζητούν οι άνθρωποι αυτοί νέα άδεια στην περίπτωση που δεν έχει ανανεωθεί η προηγούμενη και να καταργηθούν τα άρθρα τα οποία είναι περιοριστικά και τα οποία αφορούν την προστασία εσωτερικά στις χώρες προέλευσης ή και επιτόπου. Στην περίπτωση που υπάρχει φόβος δίωξης ή όπου η επικουρική προστασία διωξη η οπου ή βασίζεται σε γεγονότα τα οποία επήλθαν μετά από την αναχώρηση των ενδιαφερομένων από την χώρα προέλευσης. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μου έστειλε η συνάδελφος. Ελπίζω να μην να, στα όσα ήθελε να πει. Πρόεδρος, του Βέλτ, αντικαθέτει την ε, κυρία Μενάσο, ε, της δίνω το λόγο. Ναι, η Αγγέλικα Μίλναρ είναι σε άλλη συνεδρίαση και ζητάει συγγνώμη και θα σας διαβάσω σύντομα ε, κάποια σημεία που ήθελε να θέσει υπόψη τη εισηγήτριας. Ως και ότι η θεωρώ, λέει, ότι η αναθεώρηση του κοινού συστήματος ασύλου θα πρέπει να βασίζεται στη γνήσια αλληλεγγύη, ακόμα και στον επιμερισμό ε, των ε, ευθυνών. Έχω κάνει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή μαζί με το σχέδιο έκθεσης τι στόχο έχουν τροπολογίες, την περαιτέρω εναρμόνιση πρώτον των δύο καθεστώτων, ε, γιατί τη ε, επικορική προστασία ε, τους πρόσφυγες. Επίσης, η πρόταση ε, του Δουβλίνου για την, τον ορισμό της οικογένειας, μέτρα προστασίας σε περίπτωση που μια τρίτη χώρα μπορεί να ε, προστατεύει ε, με κάποιο μόνιμο χαρακτήρα και ουσιαστικά επίσης να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να επιλέγουν το καθεστώς. Και να πω και κάτι προσωπικό, όχι αυτό που λέει η κυρία Μιλνέρα, απαντώντας στον κύριο Χαλάχο. Εάν θέλετε να ενσωματώνονται οι άνθρωποι. Αν δεν τους δώσετε μια προοπτική μόνιμης διαβίωσης, για ποιο λόγο να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Δεύτερον, τα σχόλια που κάνετε, τι υπονοούν. Ότι οι πρόσφυγες και εκείνοι που ζητούν άσυλο και είναι ένοχοι για κακοποίηση παιδιών, για βιασμούς και βέβαια φυσικά και θα πρέπει να τιμωρούνται. Αυτό ισχύει για όλους. Δηλαδή τι θα πρέπει να ε, τιμωρούνται περισσότερο ή είναι πιο εγκληματίες επειδή είναι πρόσφυγες. Αυτό είναι πάρα πολύ επιθετικό, είναι τελείως αβάσιμο. Εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς που έχουν τέτοιες απόψεις και απόψεις που δεν συμμερίζομαι, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων περί γυναικών. Άλλο η ενσωμάτωση, άλλο η ένταξη και άλλο η αφομοίωση. Ε, και εγώ θα ρωτούσα και με ποια στάνταρτ. Και όλοι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση που αυτό σημαίνει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Λάμπερτ από του Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και την εισηγήτρια και εμεί πιστεύουμε ότι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Γι' αυτό και δεν είναι τροπολογίε όπου συμφωνούμε με την εισηγήτρια. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε κάνει τροπολογίες για όλα τα θέματα. Εκτός αν θέλουμε να επισημάνουμε κάτι για να σημειώσουμε ιδιαίτερα. Το έχω ξαναπεί, ε, θα πρέπει η οδηγία να γίνει κανονισμός ή όχι. Ακούμε διάφορους ισχυρισμούς για ενδεχόμενες επιπτώσεις αν γίνει το κείμενο κανονισμός. Αυτά είναι υπερβολικά για να το πω έτσι με τριοπαθώς. Και ορισμένοι προωθούν ε, χαλάρωση των κανόνων που Θα τα ξαναδούμε αυτά ε, όταν θα έχουμε τις προτάσεις των κρατών μελών. Κάτι που υποστηρίξαμε εμείς, οι πράσινοι, και σε τροπολογίες προωθούμε είναι να αφαιρεθούν οι αναφορές στις δευτερογενείς μετακινήσεις. Εδώ πρόκειται για μια νομοθεσία ε, που έχει να κάνει με τις απαιτήσει για την αναγνώριση ε, του τρόπου με τον οποίο χορηγείται το καθεστώς ε, του πρόσφυγα ή εκείνου που δικαιούται προστασία. Δεν έχει θέση εδώ λοιπόν η δευτερογενής μετακίνηση. επίσης την εσωτερική προστασία θέλουμε να ε, βγάλουμε. Για μας η επαρκής ε, προστασία, η ικανοποιητική προστασία των πολιτών είναι ζήτημα του κράτους. Και δεν θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να εκχωρηθεί για να το ε, ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιος τρίτος. Αυτό είναι ένα κρατικό δικαίωμα και δεν συμφωνούμε. Είναι η πρώτη ευκαιρία που έχει το Κοινοβούλιο με όρους νομοθετικούς να αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα και πραγματικά θα μας ενδιαφέρει να γίνει. Γιατί δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι από τα όσα ακούμε. Δεν έχουμε ακούσει έγκυρα επιχειρήματα για να διατηρηθεί. Επίση, συμφωνούμε πάρα πολύ με την ενοποίηση κατά κάποιο τρόπο των δύο καθεστώτων εκείνων που δικαιούνται επικορική προστασία και ε, ε, εκείνων που χαρακτηρίζονται πρόσφυγες. Δεν θα πρέπει όμως να υποχρεώνουμε τα κράτη-μέλη ε, συνεχώς να αναθεωρούν ή να επανεξετάζουν το καθεστώς. Αυτό πέρα από ένα γραφειοκρατικό φόρτο σημαίνει και υπονόμευση οποιασδήποτε εξασφάλισης των προσφύγων. Και σίγουρα δεν τους ε, παροτρύνει να εντάσσονται στις κοινωνίες όπως ακούσαμε. Και για πολλούς πρόσφυγες ε, ε, ε αυτό σημαίνει ότι θα ζουν έξω μακριά από τη χώρα τους. Ήμουν τις προάλλες στο Πακιστάν και είδα πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που τους λένε ότι δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω την επόμενη 30 ετία. Δηλαδή, όταν έχει κάποιο ένα τέτοιο χρονικό ορίζοντα και δεν μπορεί να ενσωματωθεί, εκτό από άνθρωπο, είναι και αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει λοιπόν να συμπληρώσουμε αυτά τα δικαθιστότητα, να τα ενοποιήσουμε, και... αλλά δεν πιστεύουμε ε, ότι οι ανάγκε ενό ανθρωπού είναι διαφορετικέ ανάλογα με το καθεστώ του, αν χαρακτηρίζεται πρόσφυγα ή ε, ε, έχουν ανάγκη επικουρική προστασία. την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν αναθεωρήθηκε τελευταία φορά. Επίσης, για την αμοιβαία αναγνώριση συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε ότι τα μέτρα ενσωμάτωσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Αν γίνουν υποχρεωτικά, θα πρέπει να υπάρχουν κιόλα. Γιατί σε, κράτη, μέλη, δεν μπορούμε να τα υποχρεώνουμε να ε, εξασφαλίζουν κάποια δικαιώματα σε πρόσφυγες τα οποία δεν υφίστανται. για τη χρηματοδότηση. Θέλουμε οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση για το άσυλο και τη μετανάστευση. Γιατί κάποια κράτη-μέλη έχουν ορθώσει άχρηστα εμπόδια στην πρόσβαση των ΟΤΑ ε, στη χρηματοδότηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντική ε, νομοθεσία αυτή ανεξαρτήτως του τελικού καθεστώτος και πραγματικά χαιρόμαστε που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει σκιώδηση από την ευθύτη. Έχουμε τρία, τρεις βουλευτές που ζήτησαν τον λόγο. Και μετά θα δώσω βέβαια τον λόγο στην Επιτροπή για να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μερική διάταξη, λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο αυτό το ενημερώνω. Το λέω για να ενημερώσω του κύριε Μετσόλα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Τάνια, την Αλισάνδρα και τους συναδελφούς που έκαναν πολλή δουλειά πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Ε, με αφορμή αυτά τα οποία είπε η Αλεσάνδρα να επαναλάβω και να επιβεβαιώσω ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει την πρόταση που αφορά ακριβώ την ε, εξάλληψη, την ε, μείωση των διοικητικών εμποδίων κάθε φορά που κάποιο ζητάει διεθνή προστασία. Χρειαζόμαστε μια πιο ενιαία διαδικασία ακριβώς για να μην έχουν κίνητρα οι πρόσφυγες να ζητούν διεθνή προστασία σε πάνω από ένα κράτο μέλος. Για τις δευτερογενείς ε, μετακινήσεις καταλαβαίνω αυτό που είπε η συνάδελφος, αλλά κάποια στιγμή όταν θα συζητάμε τα περί του κεκτημένου στον τομέα Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και κράτη-μέλη τα οποία κρύβονται πίσω από τις δευτερογενείς αυτές ροές για να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, είπαμε υπάρχει το φαινόμενο της ε, επιλογής χώρας υποβολής αιτήσεως γιατί διαφέρουν ακριβώς οι χώρες μεταξύ τους, διαφέρουν οι συνθήκες από χώρα σε χώρα. Αυτό, ναι, να το λάβουμε υπόψη μας εννοείται. Μπορεί να χρειαστούν πολλές συζητήσεις για το ποιες είναι οι επιπτώσεις, αλλά να δούμε τι συμβαίνει, τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη, αφού τους χορηγηθεί προστασία στο κρατομέλος Α. Και τι πρέπει να κάνουμε με τις επιπτώσεις αυτές. σίγουρα κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Συμφωνούμε επίσης ότι όλοι οι ετούντες για διεθνή προστασία πρέπει να έχουν την ευκαιρία μιας ταχείας εξέτασης της αιτησής τους. Τα κρατη στα οποία οι άνθρωποι αυτοί είναι επιλέξιμοι, πρέπει να τους βοηθούν και παράλληλα όμως να υπάρχει και μια αποτελεσματική διαδικασία επιστροφής. Να μην φτάσουμε, να μην φτάνουμε στο σημείο κάποιοι να ζουν χρόνια ή και δεκαετίες ε, μέχρι να ε, δοθεί μια τελική λύση και να έχουμε θέματα ενσωμάτωσης της τοπική κοινωνία. Μπίρκετ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζήπελ. Καταρχάς, όταν μιλούμε για επικορικές μάλλον για δευτερογενείς μετακινήσεις, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το ισχύον σύστημα ασύλου σημαίνει ότι δύο-τρεις χώρες θα είναι υποψήφιες, μάλλον αρμόδιες, υπεύθυνε να ε, διαχειρίζονται ε, όλο το άσυλο και τη μετανάστευση, η Ελλάδα και η Ιταλία, γιατί έχουμε το σύστημα του Δουβλίνου ε, που ορίζει ότι οι χώρες που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση αυτού του συστήματος είναι χώρες πρώτης υποδοχής. Αυτό είναι τελείως άδικο. Αφήστε που δεν είναι και αλληλέγγυο. Και όταν μιλούμε για δευτερογενείς μετακινήσεις, εκπλήσωμαι που ακούω ότι υπάρχει δυνατότητα να ζητάει κανείς άσυλο σε διάφορα κράτη-μέλη. Γιατί εγώ θεωρούσα ότι για να ε, αποφύγουμε αυτό έχουμε το σύστημα Eurodac, δηλαδή παίρνουμε δακτυλικά αποτυπώματα. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο λόγο διαφερομένο έχει ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα. Ε, Προφανώ δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Μήπω θα πρέπει να βελτιώσουμε τα συστήματα που διαθέτουμε αντί να αναζητούμε ε, άλλα οπισθοδρομικά μέτρα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Για την προστασία εκείνων που έχουν καθεστώς πρόσφυγα και άσυλο. Θα πρέπει να είναι πάντα προσωρινή. Ακούμε. Έχουμε μια εμπειρία, ιδιαίτερα στη Γερμανία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποδεχθεί πολλούς πρόσφυγες. Και αν λέτε από την αρχή στον κόσμο ότι ωραία σε προστατεύω, αλλά για λίγα χρόνια μόνο, τότε εκείνο γιατί να κάνει, να πει στον κόπο να ενταχθεί στην κοινωνία και να ακολουθήσει τους κανόνες. Αν του πούμε ότι σε προστατεύω ένα χρόνο μετά θα φύγεις. Εγώ τι κίνητρο έχω να ακολουθήσω τους κανόνες. Για να έχουμε τουλάχιστον την ευκαιρία να παραμένουν οι πρόσφυγες στη χώρα που ζητούν άσυλο και το λαμβάνουν. Ε, αυτό τους βοηθάει και στην εσωμάτωση. Και όταν οι άνθρωποι αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους λόγω πολέμου, έχουμε ζήσει ότι επιστρέφουν μετά τον πόλεμο. Κοιτάξτε μας τι γίνεται στη Συρία. Ο πόλεμος τώρα διανύει το έκτο έτος του. Και εκείνοι που χρειάστηκε και αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους, δεν θέλουν να παραμείνουν πρόσφυγες, ούτε για έξι χρόνια, ούτε για όλη τους τη ζωή. Θέλουν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους κάπου. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά και για την κοινωνία στην οποία ζουν και συνεισφέρουν. Και θα πρέπει να το κάνω αυτό, αντί να περιμένουν απλώς να επαναπατριστούν. Και ένα τελευταίο, να απελάβνονται ε- οι εγκληματίες, οι Αυτό με ανησυχεί, γιατί χρειάζεται δίωξη, χρειάζεται δικαστήριο και χρειάζεται δικαστική απόφαση και κύρωση όταν κάποιος εγκληματεί. Εάν τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό καθεστώς για μια ομάδα ανθρώπων που ζει στις χώρες μας, τι θα σημαίνει αυτό για το δικαστικό σύστημα ε, μακροπρόθεσμα. Εάν για την ίδια αξιόπινη πράξη έχουμε διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει ε, κάποιος. Τώρα έχουμε του πρόσφυγες. Η επόμενη ομάδα που θα έχει δικού κανόνε γιατί δεν μα αρέσει ποια θα είναι. Υπάρχει το κράτο δικαίου, υπάρχουν κανόνε που ισχύουν για όλου και ε, έτσι αντιμετωπίζονται ε, όσοι παραβαίνουν τον νόμο, είτε είναι Γάλλοι, Γερμανοί, Πολωνοί, Ρουμάνοι, Σύριοι, οτιδήποτε άλλο. Όλε οι εθνικότητε έχουμε του κανόνε δικαιοσύνη, οι οποίοι ισχύουν και θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλου. Ευχαριστώ. Thank you very much. ευχαριστώ. Ο κύριος Τσεχόφσκι έχει το λόγο. Děkuji. Krásně vyslovujete mé jméno. Tak eh, já bych... Ευχαριστώ. Έχω κάποια σχόλια. Ευχαριστώ την εισηγητρία. Το θέμα δεν είναι απλό. Και το λέω αυτό πραγματικά με θαυμασμό για το έργο των συναδέλφων. Τάνια, ελπίζω ότι θα συμφωνήσεις με κάποια από τα σχολιά μου, γιατί έχω ταξιδέψει και έχω επισκεφθεί στρατόπεδα και εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων. Ε, πρόεδρε, λοιπόν, επιτρέψτε μου Θα χρειαστώ μερικά λεπτά, λοιπόν, για τον κανονισμό. Καταρχάς, τον συνέκρινα με τον 109, ε, με τον προηγούμενο, με την οδηγία μάλλον, 25 Νοεμβρίου του 2003. Δεν βλέπω πολλές διαφορές, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές όσον αφορά το, την μεταχείριση των οικογενειών, αλλά εν γέννη κανονισμός όσο έχει έτσι όπως ε, επαναδιατυπώθηκε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μεγάλες διαφορές. Πάντως δεν κάναμε και κάτι από αυτούς που περίμεναν κάτι περισσότερο από εμάς. Όσον αφορά τις συστάσεις, κάποιες είναι σωστές θα έλεγα. Όμως, Τανία, πρέπει να δοθεί μια γενική κατεύθυνση, να υπάρχει ένα κοινό θέμα που να, να διέπει την προσέγγισή μας των προσφύγων, των οικογενειών κλπ. Από έτσι όπως βλέπω τα πράγματα τουλάχιστον, είναι δύσκολο να ορίσουμε το μέλος της οικογένειας. Ας πούμε, ένας αδελφός είναι μέλος της οικογένειας, δικαιούται προστασίας. Μήπως έτσι ενθαρρύνουμε και άλλους να έρθουν στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ότι σοβεί μια κρίση. Μετά στο άρθρο 16.1 γάμα αλφα Βλέπω εδώ ότι διευρύνουμε το πλήθος των ανθρώπων που δικαιούνται επικουρικής προστασίας. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη υποφέρει από μαζική εισρωή ανθρώπων. Εδώ τι κάνουμε, διευρύνουμε τον ορισμό Αυτόν που δικαιούν επικουρική προστασία. Φοβούμαι ότι αυτό δεν συνάδει με τον τρέχοντα ορισμό της διεθνούς προστασία. έτσι πως το διαβάζω εδώ. Και δεν είναι καν θέμα το οποίο αποσχολεί άλλε χώρε διεθνώ θα έλεγα. Εδώ θεσπίζουμε μια ε, πολύ μεγάλη αλλαγή. Και κάτι άλλο, Προσωπικώς δεν είμαι υπέρ της εναρμόνισης των διαρκειών ισχύω των διών διαμονής για όσους έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες και που απολαύουν διεθνούς προστασίας. Θεωρώ, δηλαδή, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να το ορίζουν αυτό κατά την κρίση τους. Και τέλος, η πορείδος προσαρμογής θα μπορούσε να περιοριστεί στους τρεις μήνες κάλλιστα. Το λέω αυτό διότι τέτοιε αλλαγέ, μεγάλη εμβέλεια, ιδιαίτερα ενόσο εκκρεμούν αποφάσεις δικαστηρίων, που μπορεί να ληφθούν σε ένα χρόνο από τώρα, ή λιγότερο ή περισσότερο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Μια περίοδος δύο ετών θα ήταν απόλυτα λογική. Α δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει λόγος ε, να βιαστούμε προκειμένου. Η σημερινή διαδικασία, η τρέχουσα διαδικασία χορήγηση ασύλου, νομίζω λειτουργεί. Γιατί να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Θα ήταν άτοπο. Επίσης, η Σόφη είπε προς τους συντηρητικούς συναδέλφους κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι στο πλαίσιο του ασύλου πρέπει κανείς να σέβεται τους κανόνες και τον τρόπο σκέψης του κάθε κράτους μέλους. Σύμφωνα απολύτως. Όταν λέμε λοιπόν ενιαίο, ενοποιημένο, να προσέχουμε. Εγώ πήγα σε ένα στρατόπεδο προχθές στην ε, Τσεχία στην πόλη Μπάλκοβα. Μπάλκοβα είναι και το όνομα ε, αυτού του χώρου συγκέντρωσης. Έχουμε εκεί ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν την απόφαση με την οποία είτε θα γίνουν αποδεκτοί είτε θα χρειαστεί να φύγουν. Είδα και εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι ε, απλώς είχαν παραβεί κάποιους νόμους, κάποιες διατάξεις της Τσεχίας. Είδα επίση ανθρώπους να προσέρχονται με παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Κάποιοι από αυτούς, ε, δεν λέω, είχαν ε, εμπλακεί σε εγκληματικές δραστηριότητες, ε, μπορεί ναρκωτικών, ακόμα και με οργανωμένες συμμορίες, οι οποίοι όμως είχαν ζήσει ήδη αρκετά χρόνια στην Τσεχία και οι οποίοι είχαν λάβει επεκτάσεις των αδειών διαμονής τους. Θέλω πω ότι είχε ανανεωθεί η άδειά τους, η άδεια παραμονής, παρά το γεγονό ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζονταν πλέον ειδική προστασία. Να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση Θυμίζω ότι η Τσεχία αρνήθηκε να συζητήσει, να δώσει καν το δικαίωμα σε ετούντε να υποβάλουν αίτηση, ούτε έδωσε τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασία. Πολλές φορές ε, μια διαδικασία θέλει τρία-τέσσερα χρόνια, μια διαδικασία έκδοση για παράδειγμα και πολλές φορές ε, κακές συνθήκες. Λοιπόν, ευχαριστώ για, για την κατανόησή σας. Ε, συνήθως τελειώσω ένα λεπτό, αλλά ε, αυτή τη φορά χρειάστηκε να τα πολύ πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά έπρεπε να τα πω. Κύριος Λέναρς. Uh, uh, ευχαριστώ την Τάνια για την εργασία της, γιατί θέλει να έχει μία προοδευτική προσέγγιση. Δεν ξέρω κατά πόσο το επιτυγχάνουν οι 800 τροπολογίες, αλλά πάση περιπτώσει θα μας απασχολήσει σύντοχρον. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μόνο μέτρα ε, θετικής ενσωμάτωσης. Νομίζω ότι χρειάζομαστε και θετικά αλλά και κυρωτικά μέτρα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ε, παρέχουν αυτή την προστασία σε όσους τη ζητούν, αλλά θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη ότι δεν έχουμε μια Ευρώπη à la carte, όπου ο καθένας αποφασίζει προς τα που θα κινηθεί. Και δεν νομίζω ότι μόνο τα θετικά μέτρα ε, θα είναι πραγματικά ανταποδοτικά. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Σίπελ, ότι φυσικά ε, έχουμε και τη Eurodac για να μην έχουμε δευτερογενείς ε, μετακινήσεις. Αυτή τη στιγμή μας απασχολεί η Eurodac και μέχρι τώρα δεν γίνεται καμία αναφορά στις δευτερογενείς μετακινήσεις στο κείμενο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε λοιπόν μία υποστήριξη και ως προς τις ε, αλλαγές στη Eurodac. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπήρχε και ένα τελευταίο αίτημα από τη Σόφη Ιντβέλτ ε, για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Συμφωνώ με την κυρία Ζίπελ ότι το θέμα της δευτερογενούς μετακίνησης έχει συζητηθεί σε άλλα φόρα και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν κίνητρα και φυσικά να υπάρχει και ένα κυρωτικό πλαίσιο τη στιγμή που θα πρέπει να ε, ε, επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Χόφτλικ μίλησε για τις αξίες, για αξίες δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να συμμερίζονται τις δικές σας αξίες, όχι τις δικές μου. Αλλά θα πρέπει να τηρούν το νόμο. Άκουσα πολλές δηλώσεις από αυτούς που είναι κατά της μετανάστευσης αλλά και ζητάνε γιατί πρέπει να προσερτεριστούν τις αξίες μας. Αλλά αυτοί που τα λένε αυτά Ξέρουμε τι αξίες έχουν σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα ως προς τους ομοφιλόφιλους, ΛΟΑΔ και ούτω καθεξής. Ωραία. Ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ καλωσορίζουμε τις τροπολογίες, ιδιαίτερα εκείνες που ενισχύουν, ε, ενισχύουν τις προτάσεις της Επιτροπής. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σας, να το βάλετε λίγο πιο κοντά. Καλωσορίζουμε, όπως είπα, την έλευση των τροπολογιών, ιδιαίτερα εκείνες που ενισχύουν τους στόχους της ε, πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που έχει σημασία είναι ιδιαίτερα τα μέτρα ενσωμάτωσης που προβάλλονται από τα κράτη-μέλη, καθώς και τους ανηλίκους, ιδιαίτερα όσον αφορά την κυδαιμονία τους. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τη θέση των περιβαλλοντικών μεταναστών. Δεν θα πρέπει να υπάρχει έλλειψη προστασία, προστασίας τους. Επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα στόχο που ήταν ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της ε, πρότασης σε σχέση ε, με τη χορήγηση ασύλου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ενιαίο σύστημα και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει χρήση της εναλλακτικής, της εσωτερικής προστασίας που είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε λόγος και για την προοπτική ενσωμάτωσης. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ένα από τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα παραμονής ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας. Εάν υπάρχει λόγος ενσωμάτωσης μέσα στα πλαίσια της νόμιμης μετανάστευσης ως προς την απόσυρση του καθεστώτος, γιατί μιλήσαμε για ε, στοιχεία που αποδεικνύουν ε, εγκληματικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Η Επιτροπή κωδικοποιεί την ομολογία επί του θέματος. Δεν εισαγάγει νέα στοιχεία. Και ως προς τις δευτερογενείς μετακινήσεις, η πρόταση αυτή δεν ε, προβλέπει νέους ε, όρους, απλώς αντικατοπτρίζει τον κανονισμό του Δουβλίνου από πλευράς δικαιούχων. Δηλαδή, ο δικαιούχος θα πρέπει να παραμείνει στο κράτος μέλος όπου την χάνει προστασίας, δηλαδή δεν πρέπει να ε, μεταβεί σε ένα άλλο κράτος μέρος, μέλος χωρίς ε, να υπάρχει λόγος. Μπορεί δηλαδή δυνάμει των κανόνων του Σέγγεν, αλλά δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να επικροτήσουμε αυτή τη μετακίνηση. Ευχαριστούμε. Η κυρία και τι ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνει αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Ε, λίγο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Έχουμε δύο θέματα από κοινού, το Φορέα Ευρωπαϊκών Εθνιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Περιμένουμε για λίγα λεπτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, γι' αυτό ας διακόψουμε για δύο-τρία λεπτά. Αλλά μην πάτε και πολύ μακριά. Uh, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμα καθοδόν, φαντάζομαι εντός του κτηρίου, αλλά δεν θέλω να σας αφήσω να περιμένετε ακόμα περισσότερο. Το Σεπτέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για τον ΜΠΕΡΕΚ και τον ε, κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ε, αναδιατύπωση τέσσερων οδηγιών είναι αυτή. Ε, επί της ουσίας αρμόδια για τα δύο είναι η Επιτροπή Ήτρε, εμεί γνωμοδοτούμε. Τα θέματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους στενά και αποφάσισαν ε, οι συγητής και οι συντάκτες να τα συζητήσουμε μαζί. Και τον κώδικα λοιπόν και τον Μπέρεκ. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Πέτερσεν και θα μας παρουσιάσει τώρα το σχέδιο γνωμοδοτήσεών του και τις δύο γνωμοδοτήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν φτάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία. Ιδιαίτερα το σε... Μανουέλ και τον Γιώργη για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και την πολύτιμη βοήθειά τους για τα δύο αυτά θέματα. Είπατε ότι είμαι εγώ συντάκτης και για τις δύο γνωμοδοτήσεις. Είχα το προνόμιο να προσπαθήσω να τροποποιήσω το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ε, που είναι πολύ σημαντικά για μας, διαφάνεια, αξιοπιστία, προστασία ε, της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Για τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καλωσορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κανονιστικό. Ε, επιτυχής όμως ε, ε, υλοποίηση και εκτέλεση θα πρέπει να εγγυάται την πολυφωνία, την πολιτιστική ε, ποικιλία την προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής, προστασία των καταναλωτών κλπ. Γι' αυτό προς την κατεύθυνση αυτή πηγαίνουν οι προτάσεις μου για τροποποίηση του κειμένου και ταυτόχρονα λαμβάνουμε υπόψη και την επικείμενη αναθεώρηση οδηγίας για την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το λεγόμενο e-privacy και την προστασία ε, τον αντίστοιχο κανονισμό. Άρα προσπάθησα, όπως βλέπετε, να εξασφαλίσω κανόνες ίσους για ε, όλους τους ε, παρόχους ε, υπηρεσιών για τις διαπροσωπικές επικοινωνίες και ταυτόχρονα εξασφαλίσουμε κοινά πρότυπα για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών προστατεύοντας πάντα τον τελικό χρήστη και την ιδιωτική του ζωή. Όπως μπορεί να θυμάστε πρόσφατα εγκρίναμε μια πρωτοβουλία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και πώς αυτά συνδέονται με τα big data. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής μας θα πρέπει και εμείς ε, να προωθούμε ε, την κρυπτογράφηση ε, για να είναι ασφαλής η πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες. Χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια που θα αποδυνάμωναν την ασφάλεια των δικτύων μας. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα επίσης προτείνουμε να δημιουργηθεί ένας φορέας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Μπέρεκ. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα. Για να ενημερωθεί το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ το κάνουμε αυτό για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ότι είναι σε θέση οι ρυθμιστικές αρχές να επιτελούν το έργο που περιμένουμε από αυτές. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχυθούν λοιπόν οι ε, αρμοδιότητες του Μπέρεκ, που είναι ο ενιαίος φορέας. Θα πρέπει και εκεί να λαμβάνονται υπόψη θεμελιώδεις αρχές και ε, οι αξίες, όπως αναγνωρίζονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει ο Μπέρεκ να είναι ένας οργανισμός ισχυρός, ανεξάρτητος, διαφανής και να ανταποκρίνεται στο έργο του που είναι η ε, αποτελεσματική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια παντού. Αυτό ισχύει για τους παρόχους, για τους χρήστες και για τη λειτουργία του Μπέρεκ φυσικά. Περιμένω να ακούσω ε, τις προτάσεις σας ε, και τα σχόλιά σας με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Και πάντα οι πόρτες του γραφείου μου θα είναι ανοιχτές. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ο λόγο του οι εισηγητέ, που είναι παρόντε τουλάχιστον κύριο Σκρίπεκ, παρακαλώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Έκανε πολλή δουλειά. Θέλω να υποστηρίξω το κείμενο, για να υποστηρίξουμε το τομέα της τεχνολογίας, για να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε μπροστά μας ευκαιρίες, όμως και προκλήσεις όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένας κανονισμός τι κάνει, συγκεράζει ακριβώ αυτά τα δύο, τις ανάγκες ε, εποπτείας από τη μια μεριά με την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων από την άλλη. Είμαι υπέρ λοιπόν της ανεξάρτητης ε, εμπειρογνωμοσύνης του Μπέρεκ. Όμως δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτό δεν θα μας βοηθήσει όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη, θέση χωρίς την γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εθνικοί οργανισμοί, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη όπως το κάνουν άλλωστε και σήμερα. Αν λοιπόν το σύστημα λειτουργεί, γιατί να το χαλάσουμε, γιατί να το αλλάξουμε. Αυτή είναι η θέση μου. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλον σκιώδη βουλευτή που να θέλει τον λόγο. Δεν εγώ τις ευκαιρίες ως ε, σκιώδη εισηγητής για να πω δύο λόγια για το σχέδιο γνωμοδότησης. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι καλή σύμβουλη προς την Ήτρα, την Επιτροπή Ήτρα και νομίζω ότι καλώς υπογραμμίζουμε την ανάγκη κρυπτογράφησης καθ' όλο το μήκος της διδρομής ενός μηνύματος και μάλιστα θα ζητούσα και κάτι περισσότερο. Μήπως ε, έχουμε την ευκαιρία εδώ, μια που κάνουμε μεταρρυθμίσεις μια φορά στα 10 χρόνια, μήπως ε, θα έπρεπε η κρυπτογράφηση, η ηλεκτρονική κρυπτογράφηση, είναι υποχρεωτική καθόλου το μήκος της διαδρομή ενό μηνύματος, μιας επικοινωνία. Αυτά, αυτή είναι μια σκέψη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από εδώ και πέρα. Ε, αν δεν θέλει τον λόγο κάποιο άλλο, ε, δίνω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και θέλετε τον λόγο ξανά. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά τα γραφή μας είναι πολύ μακριά από το Κοινοβούλιο. Είδαμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια στον εισηγήτη. Ευχαριστώ και για τα σχόλιά σα σήμερα. Άλλε επιτροπέ έχουν υποβάλει παρομοίε τροπολογίε Θα συνεργαστούμε βεβαίω. και θα κάνουμε πανδυνατόν για να σωματώσουμε τις παρατηρήσει του Κοινοβουλίου στο τελικό κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστώ την Κομισιόν. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, φτάμε και εμείς γιατί ξεκίνησαμε λίγο νωρίτερα, μη ζητάτε συγγνώμη. Ο λόγος των κ. Πέτρεσεν ως συγγητή. Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρόθεση της κρυπτογράφησης, ακόμα και την πρόταση να γίνει και υποχρεωτική. Να το συζητήσουμε, να δούμε τι επιπτώσεις θα είχε κάτι τέτοιο. Είμαι θερικά διακείμενος, καταρχήν τουλάχιστον, να το δούμε, να το συζητήσουμε. Πώς τον κύριο Κρύπε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω γιατί διαφωνείτε για την δημιουργία ενός νέου οργανισμού. Η ανάγκη μας υπάρχει, πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά Καταλαβαίνω, δικαιούστε να διαφωνείτε, να λέτε ότι δεν είναι ανάγκη. Όμως, όμως, με βάση το διαθέσιμο υλικό της προτάσεις και τα στοιχεία που έχουμε στη διαθέσή μας, πιστεύω ότι είναι δικαιολογημένη η αποφασή μας. Καλώς, λοιπόν, δημιουργούμε ένα νέο οργανισμό. Με αυτά, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Όπως είπα, επικοινωνήστε μαζί μου οποτεδήποτε θέλετε εάν θέλετε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Να ενημερώσω την Ομίγυρη ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι η 3η Μαΐου, 10 το πρωί. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, οπότε να προετοιμαστείτε παρακαλώ καταλήλως. Και μην ξεχνάτε ότι οι τροπολογίες για το κωδικοποιημένο μέρος πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολόγηση βάσει του 105. Λοιπόν, προετοιμαστείτε προσεκτικά όσον αφορά τις τροπολογίες και να βεβαιωθείτε ότι είναι σύμφωνες με τον κανονισμό, αλλιώς δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτά. Είχα μια ωραία ζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από δραστηριότητε ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο για τη σχετική οδηγία. Προχώρησε ο τριμερή διάλογος. Ο επόμενος είναι στις 10 Μαΐου. Η κυρία Σαρσεντίνη είναι συνεισηγητρία από τους φιλελευθέρους ε, θα μας ενημέρωνε από τους πρασίνους που ε, ε, δεν μπόρεσε να, είναι εδώ θα μας ενημέρωνε λοιπόν πέρασε ένας χρόνος από τις διαρροές των Panama Papers αυτή και άλλες εξελίξεις που γραμμίζουν την ανάγκη διαφάνειας όσον αφορά τα θέματα του ξεπλήματος και της φοροδιαφυγής πρέπει να απαγορεύσουμε την απόκρυψη εσόδων στους εγκληματίες. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις τρίτες χώρες και δι τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δύο τριμερείς διάλογοι έγιναν ως σήμερα για την ε, πρόληψη του ξεπλήματος. Ε, ο επόμενο είναι τον Μάιο. Προκύπτει σαφώ από τις διαπραγματεύσεις ότι όλοι θεωρούμε σημαντικό το να καταλήξουμε σε ένα αυστηρό πλαίσιο για την απαγόρευση της ε, φόρο του ξεπλήματος και τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας. Συζητήσαμε κατά πρώτον τα Μητρώα όσον αφορά τους ε, πραγματικούς δικαιούχους, ε, τους πραγματικούς μετόχους διαφορών επιχειρήσεων. Τονίσαμε επίσης την σημασία πρόσβαση σε αυτά τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων, δηλαδή των μετοχών ε, των επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια τα οποία θα μπορούσαν να εξυπήσουν οι εγκληματίες. Σύμφωνα με την ε, θα καταθέσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου στον επόμενο γύρο. Όπως είπε η κυρία Σαρζεντίνη, ο επόμενο γύρος είναι 10 Μαΐου του τριμερού διαλόγου και δεν ξέρω αν η Κομισιόν έχει να πει κάτι προκειμένου δεν το θεωρώ όμω. απαραίτητο καθώ έκανα μια απλή ενημέρωση. Τώρα, διακόπτουμε ως τις ε, ψηφοφορίες που είναι στις 11 και 40. Έχετε λίγα λεπτά στη διάθεση σας λοιπόν να πάρετε στα γρήγορα ένα καφέ. Ευχαριστώ. Just to repeat, meeting is suspended until... Να παραλάβω ότι έχουμε διακόψει ως τις 11 και 40.

Okay. Okay, dear... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, I ask you to sit down, please. Καθίστε παρακαλώ. We would like to start ψηφοφορίες και θα θέλαμε να αρχίσουμε. And we will start... Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειε κυκλοφορία οχημάτων στην Κροατία. Εισηγητής είναι ο Κλοντ Μωράης, τον οποίο και αντικαθιστώ σήμερα. Ψηφίζουμε. Είναι απλοποιημένη η διαδικασία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ψηφοφορία Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας. Παραλίγο να πω το Ηνωμένο Βασίλειο. για συμπληρωματικού κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020. Εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεσης, ψηφίζουμε, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Ευχαριστούμε τον εισηγητή τον κύριο Σεχόφσκι. Επόμενη ψηφοφορία. Πολιτέ πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2018-2022. Η είναι η κυρία Αγγέλικα Καμίλνα. Να ψηφίσουμε και πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τις ψηφορίες. Ε, πρόκειται για έγκριση του Κοινοβουλίου. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούνατσεκ, έχω ξεχάσει την κάρτα μου ψηφοφορία. Παρακαλώ να μετράτε και εμένα. Ναι, θα το σημειώσουμε στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Καλώ, προχωρούμε. Στην επόμενη ψηφοφορία. Απαιτήσει για την υποδοχή των ετούντων διεθνή προστασία. Αναδιατύπωση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Νετφέλτ. Έχουμε μια τεχνική διόρθωση να ανακοινώσουμε. Η πρώτη πρόταση της δεύτερης παραγράφου στην συμβαστική 21 μετά το effectively λέει και ε, σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω από 20. Είναι μια τεχνική διόρθωση αυτή. Συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ την εισηγήτρια να λάβει το λόγο. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Ψηφίσουμε λοιπόν. Τροπολόγια 52 και 53 που είναι ταυτόσιμες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, μάλιστα πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1α. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1β. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2, αρχής ψηφοφορία. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3, αρχής ψηφοφορία. Και λίγη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, αρχής ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Επίσης, συμβαστική 5, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6, Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η τσαπολογή 207. Μόνο το δεύτερο τμήμα όμως, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ένας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7α και 7c μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολόγια 235 και 236 μαζί ταυτίζονται αυτές οι δύο αρχής ψηφοφορία. Περάσει. Απορρίπτεται το σύνολο. Τροπολογία 237 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με συμβαστική 7β αρχίζει υποφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Minus. In Α, δεν απορρίπτεται. Με την ψήφο της κυρίας Λούνατσεκ εγκρίνεται. τσεκ, φωνές από κάτω. Okay. So... Καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την ψηφοφορία για να την επαληθεύσουμε. Και η κυρία Λούνατσεκ που δεν έχει την κάρτα της. Αρχίζει η ψηφοφορία. Στο 7β. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Τώρα όμως. 27-26. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες 238 και 239. Ταυτόσιμες είναι αυτές, αρχής ψηφοφορία. και λίγη. Απορρίπτονται. Ε, θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 31. Θα Συγγνώμη, αρχίζει η 31. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 255 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9α, η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9β, η ψηφοφορία. Τώρα Απορρίπτεται. Άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 282. Αρχή πληροφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 284 αρχίζει η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. That's rejected. Amendment. Απορρίπτεται. 285 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική 10. ψηφιζουμε αρχή αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11α και 11c και 11η ε, όλα μαζί, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 11β, αρχής ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίζουμε την 311, η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 310 ψηφι με μάλλον αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11D αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. Και μία ψήφο από το ΕΛΚ, δεν το ξεχνάμε. Όχι ε, Α, μία υπεράριθμη. Λάθος, έχουμε μία παραπάνω από το ΕΛΚ. Uh, e από το ΕΛΚ ε, να βγάλει μία κάρτα. Ευχαριστώ. Ωραία. Το κλείσαμε. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε συμβιβαστική 12α και 12γ από κοινού ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 12β. Ψηφίζουμε. Πέρας Ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 357, 357 ψηφίζουμε. Και πάλι ε, μια υπεραριθμή κάρτα από το ΕΛΚ. Ωραία, τακτοποιήθηκε πέρας ψηφοφορία Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14. Ψηφίζουμε. Είναι 14 έτσι. 14. Συμβαστική. Και πάλι το ΕΛΚ έχει μια υπεράριθμη κάρτα. Ωραία. Τακτοποιήθηκε πέραση ψηφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Ψηφίζουμε. Και πάλι κάτι γίνεται. Ε, έχουμε μία παραπάνω ψήφα από το ΕΛΚ. Ωραία. Ευχαριστώ πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16α. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 16β. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17α και 17δ. Από κοινού ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται. Περνάμε στην 427. 4, 2, 7 και 428 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. της ψηφορίας. Απορρίπτεται. 429. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17β. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17γ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεστική 18 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 19 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης συμβαστική 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβαστική 22. Ψηφίζουμε. πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική 23, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική... Α, με συγχωρείτε, όχι. Ε, στην 518. Πάμε στην 518, ψηφίζουμε. Πέρας απορριπτεται 519 ψηφίζουμε. Πέρας. 520 ψηφίζουμε. Πέρας. 521 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρινέται. Συμβαστική 25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Ψηφίζουμε. πέρας εγκρίνεται τροπολογία 54 λέει ο πρόεδρος 54 λέει ο πρόεδρος πέρας απορρίπτεται 55 ψηφίζουμε Πέρας. Απορρίπτεται. 56. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 60. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 33, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 34, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35, ψηφίζουμε. Πέρας Εγκρίνεται συμβαστική 36. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 39. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική, μάλλον όχι, 97. 97 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 96 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορίας. Με την κυρία Λούνατσεκ εγκρίνεται με την ψήφο της. 98. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 99 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 100. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Όχι. 108. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 45. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 122. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 123. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Τροπολογία 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Όχι, όχι, καταπίπτει. Συμβαστική 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 49. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 135. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 137. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έμπλ 31. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Έμπλ 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμπλ 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και επίσης εγκρίνεται. Έμπλ 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. Εμπλ 2, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εμπλ 15, σε σχέση με την προσθήκη του αρχικού κειμένου για τις πρακτικές dumping. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την αρχή της έναρξης των διαπραγματεύσεων και την εντολή, τη σχετική εντολή, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. Να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Εντάξει, τα καταφέραμε συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.